Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar la reunión. Καλησπέρα σα. Αρχίζουμε με επαγγελματική συνεδρίαση τη Επιτροπή των ε, Αναφορών και καλώ ορίσατε και θα αρχίσω την ε, συνεδρίαση με κάποιε ανακοινώσει σχετικά με τα όσα είπαν το πρωί οι συντονιστέ. Ε, Έργαν τι εξή αποφάσει, κάτι το οποίο έχει να κάνει με τα όσα θα κάνουμε το Φεβρουάριο και εξή. Εγκρίθηκε το πρόγραμμα του Φεβρουαρίου και οι μέρες διατάξεις σε, σε σχέση με τα εργοστάσια στον Τάραντα τα υπόλοιπα θέματα θα πάνε σε άλλη συνεδρίαση και η 70-12 και ε, δεν θα πάει στην μέση διατάξη του Μαρτίου γιατί θα έχουμε εκλογές στην Σλοβακία και οι σχετικές αναφορές μας θα πάνε στο μέλλον. Θα αποφασίσουν το που θα το βάλουμε οι συντονιστές σε κάποια άλλη συνεδρίαση και θα μπουν σε κάποια. Η η 971 του 14, ε, η 1800 του 14 επίσης και η 2032 θα πάνε στον ε, Μάρτιο και ε, δύο που θα πάνε του 13 θα πάνε τον Απρίλιο του 2014 θα πάει ε, σε μια συνεργασία που θα συζητήσουμε τα σχετικά με την παιδική εργασία. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό το οποίο αποφάσισαν οι συντονιστέ. Πρόκειται για κάποια ε, προφορική ερώτηση κοινή με τη νομική επιτροπή για τα δικαιώματα των ανηλίκων. Επίσης πρόκειται να γίνει ένα ψήφισμα στα πλαίσια του κανονισμού εργασίας του Κοινοβουλίου. Στα πλαίσια αυτής της προφορικής ερώτησης επίσης πρόκειται να ε, ε, εντάξουμε ε, και, αυτή την, και, αυτό το ψήφισμα στα πλαίσια προφορικής ερώτησης τώρα. Είπαμε ότι το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα θα αναλάβει την έκθεση σε σχέση με τα ανθρώπινο δικαιώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, όσον αφορά την αξιολόγηση τη Επιτροπή για το πρόγραμμα εργασία τη Επιτροπή για το 2016, αποφασίσαμε, όπω προτείνει η κυρία Καμπεθόν, να στείλουμε τα σχόλιά μα ει την διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών. Σχόλια και τις πληροφορίες που θέλουμε να μας διαβάσουν. Επίσης, στην ε, διάσκεψη των συντονιστών επιβεβαιώθηκε το τι ισχύει όσον αφορά την δημοσία ακρόαση για την χάρτα των θεμελιωδών δικαιωμάτων που θα γίνει στο μέλλον. Επίσης, 15 Τρίτου ακρόαση για την ιδιότητα του Ευρωπαϊκού Πολίτη ε, επίσης είπαμε ποιες θα είναι οι προθεσμίες τόσο ώστε να αποσταλούν κάποιες προτάσεις για τις ακροάσεις αλλά και τις ε, ε, ερευνητικές αποστολές 4 Δευτέρου θα είναι η ημερομηνία και οι συντονιστές διατύπωσαν κάποιες προτάσεις για την γραπτή διαδικασία οπότε και θα αποφασίσουμε αλλά για αυτές που δεν θα απαντηθούν ε, ε, εγγράφως, είπαμε ότι θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει σε κάποια ακρόαση όπως ας πούμε για τους αναπήρους και είπαμε ότι θα κάνουμε και κάποια αποστολή στην Ευρώπη να δούμε πού είναι τα πράγματα ε, δύσκολα που υπάρχουν προβλήματα με τα δικαιώματα των ανηλίκων και των προσφύγων αλλά και των μεταναστών όλα αυτά θα διεκπαιριωθούν εγγράφως και θα ε, ληφθούν τελικές αποφάσει στην επόμενη συνάντηση των ε, συντονιστών. Επίση, η προθεσμία για να μου πείτε ποιοι ενδιαφέρονται για την αποστολή μα στην Ιρλανδία θα πρέπει να έχουν κοινοποιηθεί στη Γραμματεία πριν τι 16 Φεβρουαρίου. Επίση, ε, τα υπόλοιπα θέματα που ζήτησαν οι συντονιστέ πάνε για τον Φεβρουάριο. Τώρα θα ε, ε, θα πρέπει να εγκρίνετε τα πρακτικά της 12ης Νοεμβρίου και 3ης ε, Δεκεμβρίου. Αν δεν έχετε κάποια ένσταση ή κάτι άλλο να πείτε, θεωρώ ότι τα πρακτικά αυτά εγκρίνονται. Y a continuación a... Στη συνέχεια τώρα θα δούμε ποιες είναι οι σημερινές αναφορές. Έχουμε πρώτα πρώτα την αναγνώριση των υιοθετών υιοθεσιών των διασυνοριακών. Επίσης έχουμε τώρα την αναφορά 2114 του 14 και 2349 του 14 που από την Πολωνία όσον αφορά ε, τις υποσχετικές σε σχέση με το εργατικό δίκαιο και επίσης αυτού του ταξιόγραφα τα οποία ε, κλείδονται μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου. Και ο Λελούς είναι εδώ. Ωραία, καλώς ορίσατε. Έχετε το λόγο για πέντε λεφτά κύριε. Ε, witam wszystkich serdecznie. E, złożyłem tutaj petycję. Zwracam się z rząd... Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα κατέθεσα μια τέτοια αναφορά, της οποίας ο σκοπός είναι ο εξή. Να συνδεθεί αυτό με το εργασιακό δίκαιο. Το 2008 λοιπόν η ιστορία μου. Προσελήφθησα σε μια εταιρεία για παραγωγή παραθύρων ε, ως τεχνικός και μου είπαν ότι θα έπρεπε να υπογράψω μια λευκή επιταγή σε περίπτωση που θα προκαλούνταν κάποια ζημιά ε, άνω των 5.000. Παρακαλώ, μπορείτε να μιλάτε λίγο πιο αργά για να είναι δυνατόν να μεταφράσουμε αυτό το οποίο λέτε. Και στην περίπτωση αυτή, στο τέλος του έτους θα μου επιτρεφόταν η σχετική επιταγή. δεν μετά την... Ε, Έχει ένα πρόβλημα, δεν ακούγεται η μετάφραση από τους ε, διερμηνείς σε κάποιες γλώσσες. Για να προσπαθήσουμε τώρα να το διορθώσουμε. Συγγνώμη που σας διακόψαμε. Ας συνεχίσουμε. Ε, Adelante. Μάλιστα. Αυτό το γραμμάτιο λοιπόν η διαταγή θα το λαμβανά στο τέλος της σύμβαση. Αυτό δεν ε, συνέβη και αναγκάστηκα να προσαγάγω λοιπόν την εταιρεία. Η εταιρεία είχε καταστρέψει όμως, ε, είπε το σχετικό γραμμάτιο. Δεν έχω όμως οποιαδήποτε τέτοια απόδειξη, οποιαδήποτε αποτεκτικό στοιχείο ότι έχει πραγματικά καταστραφεί, ότι έχει, ε, δεν έχει πολιθεί σε κάποιους άλλους αυτό το γραμμάτιο σε κάποιον τρίτο. Το δικαστήριο λοιπόν αποφάνθηκε στο 2011 ότι σύμφωνα με το πολωνικό εργασιακό δίκαιο απαγορεύεται να θεωρηθεί ένα είδος εγγύηση το γραμμάτιο αυτό, εις διαταγή για ενδεχόμενες ζημιές που θα προκαλούσε ενδεχομένως ο εργαζόμενος. Αυτό σημαίνει ότι είναι πραγματικά αντίθετο με το νόμο το γραμμάτιο αυτό. Το άνωτο λοιπόν δικαστηρίο αποθάνθηκε ότι σε καμία διατάξη του εργασιακού δικαίου δεν προβλέπεται η έκδοση τέτοιων γραμματείων στο τομέα της νομοθεσίας. Πρόκειται για αξιόγραφα, ξέρετε. Ο εργοδότης, ο οποίος κατέχει τα γραμμάτια αυτά, θα μπορούσε να απαιτήσει την εξόφληση ε, του γραμματίου αυτού από τον εργαζόμενο και σε περίπτωση που δεν γίνει αυτή η εξόφληση πολύ απλά μπορεί να πάει στα δικαστήρια ο εργοδότης και να ζητήσει την αποπληρωμή του γραμματίου. Αυτό λοιπόν είναι μια σχετική με μια σχετικά απλή διαδικασία για τον εργοδότη και μια πάρα πολύ ε, χρονοβόρα διαδικασία για τον εργαζόμενο. Δεν δικαιολογείται δε ούτε η έκδοση ούτε το ύψος του γραμματείου για την ε, ενδεχόμενη πιθανή ζημιά. Και μπορεί να το απολύσει και σε τρίτους ε, ενδεχομένω. Και αν το αποκτήσει λοιπόν ένα τρίτο το γραμμάτιο αυτό, μπορεί να απαιτήσει ο τρίτο την αποπληρωμή του ποσού εις ολόκληρων. Δεν υπάρχει δε και καμία συγκεκριμένη διάταξη στο εργασιακό δίκαιο που δεν μπορούσε να το επιτρέψει αυτό το γεγονός. σε ό,τι αφορά μελλοντικέ αξιώσεις του εργοδότη. Σήμερα οι εργοδότες έχουν πολλές δυνατότητες. να λάμβουν αποζημιώσεις από τους εργαζόμενους σε περίπτωση πρόκλησης ζημιάς. Γιατί έχει και ηλικία ευθύνη ο εργαζόμενος. Αν όμως ο εργοδότης α, στέλνει για παράδειγμα τον εργαζόμενο για μια κατάρτιση, μπορεί να τον ασφαλίσει. Σε περίπτωση που ο και μπορεί να ασφαλιστεί και ο ίδιο εργοδότη σε περίπτωση που, για παράδειγμα, ο εργαζόμενο δεν ολοκληρώσει την εκπαίδευση. Για τα γραμμάτια, λοιπόν, πρόκειται για ένα μεγάλο πρόβλημα. Και οι επιθεωρητέ εργασία δεν έχουν ε, κάποιο συγκεκριμένο μέσο στα χέρια του για να αντιδράσουν, για να επιλύσουν το θέμα αυτό. Δεν έχουν δικαίωμα να καλέσουν καν του εργαζόμενου, του εργαζόμενου να εγκαταλείψουν τι πρακτικέ αυτέ ή να ακυρώσουν τα γραμμάτια πολύ απλά. Αυτή η εξέλιξη λοιπόν στην αγορά εργασία έχει ως συνέπεια τελικά οι εργαζόμενοι οι οποίοι πραγματικά θέλουν μια θέση εργασίας να αναγκάζονται να υπογράφουν τα γραμμάτια αυτά. Αλλά να μην αντιλαμβάνονται πλήρως την έκταση των συνεπειών. Και το φαινόμενο αυτό πραγματικά έχει πάρει μαζικές διαστάσεις. Οι εργαζόμενοι βρίσκονται τελικά μια κατάσταση, μια κατάσταση όπου την χάνουν εκμετάλλευση πολύ απλά. Ο εργοδότης δε μπορεί να προσαγάγει τον εργαζόμενο στο δικαστήριο. Και αυτό συνδέεται με υψηλό κόστο και τα γραμμάτια μπορεί να χρησιμοποιηθούν ει βάρο των εργαζομένων. Πρόκειται λοιπόν για συγκεκριμένη δράση κατά του εργαζόμενου. Γι' αυτό λοιπόν σα καλώ να απαγορευτεί αυτή η χρήση γραμματιών. Από την υπηρεσία μελετών του Κοινοβουλίου έχουμε τον κύριο Μάρκο ο οποίος έχει συγγράψει μια μελέτη όσον αφορά αυτά τα γραμμάτια λευκά και ε, λευκό και τα υπόλοιπα. Έχετε τον λόγο κύριε. Αξιότιμα μέλη, ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε σε αυτή τη συνεδρίαση. Να πω ότι εκπροσωπώ την αμερόληπτη νομική έρευνα που έκανε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ερευνητική Υπηρεσία του Κοινοβουλίου. Δεν είναι νομική όμως θέση, μόνο η νομική υπηρεσία μπορεί να το κάνει αυτό. Θα σα δώσω τρία θέματα. Πρώτα απ' όλα, εν συντομία, οι νομικές πτυχές του θέματος της ελευκό χρήσεως αυτών των επιταγών στην Πολωνία. Ποια είναι η αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ενώσης μετά, γιατί έχει δικαίωμα να κάνει κάτι η Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με το πλαίσιο των συνθήκων. Και τρίτον, συγκριτική οπτική γωνία που θα είναι με παρουσίαση της έρευνας που έκανε η υπηρεσία μας κατόπιν αιτήματος βουλευτών. So first of all, as the petitioner already... Όπως ήδη εξήγησε ο αναφέρον, αυτές οι επιταγές που έχουν ε, τα λέτρα de change στα γαλλικά είναι υποσχετικές. Ουσιαστικά, εν λευκό, διέπονται από ένα νόμο το 1936 και με πολωνικό δίκαιο μπορεί να είναι λευκές. Ο πιστωτής μπορεί να συμπληρώσει ένα ποσό. και μετά ο φιλέτης θα πρέπει να καταβάλει το ποσό. Ο πιστωτής μπορεί να μεταφέρει σε τρίτο μέρος αυτή την υποσχετική, ένα τρίτο μέρος να τη μεταβιβάσει έτη περαιτέρω και ο τελευταίος που θα πάρει αυτό το χαρτί μπορεί να ε, μηνύσει τον Φιλέτη χωρίς να υπάρχει κάποια άμεση νομική σχέση μεταξύ τους. Και έτσι ο φιλέτης, μάλιστα είναι εργαζόμενος, είναι σε δυσχερέστατη θέση, διότι ο εργαζόμενος θα πρέπει να κινηθεί και ο εργαζόμενος θα πρέπει να κάνει κάποια πράγματα, νομικά βήματα, για να μπλοκάρει την υλοποίηση αυτής υποσχετικής, αυτού του, αυτού του, αυτής επιταγής. Γιατί έχει ακολουθούνται απλή διαδικασία. Ο νόμος στην Πολωνία το καθορίζει σαφώς τι γίνεται. Τη μεταβίβαση δηλαδή δεν τη ρυθμίζει λεπτομερό στο το Δικαστήριο της χώρας ενέκρινε την χρήση αυτών των αξιογράφων την κομμουνιστική περίοδο, τη δεκαετία του 1980 ενέκρινε το θέμα αυτό το δικαστήριο και επί 30 χρόνια ενέκρινε την ανλογό πρακτική σιωπηρός. Στην υπόθεση του 2011 το δικαστήριο θεώρησε ότι αυτές οι υποσχετικές που χρησιμοποιούνται στις εργασιακές σχέσεις, δηλαδή από εργοδότη έναντι εργαζομένου, ζητώντα από τον εργαζόμενο να υπογράψει τέτοια αποσχετική εν είναι κάτι άκυρο γιατί παραβιάζει την νομοθεσία, την εργασιακή. Φαίνεται ότι αυτό το ακολουθούν και άλλα δικαστήρια, χαμηλότερα από τον νότατο. Αλλά από ανακοινώσει στον τύπο είδαμε ότι η πρακτική από εργοδότε συνεχίζεται. Να υπογραμμίσουμε. Αυτή η απόφαση του δικαστηρίου του 2011 δεν είναι δεσμευτική ως νομολογία. Το νομικό δίκαιο της Πολωνίας δεν ξέρει, δεν έχει δημιουργήσει το προηγούμενο δεσμευτικό και αυτή η απόφαση δεν δεσμεύει καν το το δικαστήριο. Η απαγόρευση της χρήσης αυτών των αξιογράφων λοιπόν στις εργασιακές σχέσεις δεν ρυθμίζεται με συγκεκριμένο τρόπο. Έτσι δε περαιτέρω, αυτή η πρακτική, ακόμα και αν υποθέσουμε ότι σύμφωνα με τον εργασιακό κώδικα είναι νόμιμη, αυτή η πρακτική είναι νόμιμη σύμφωνα με συμβάσεις απασχόλησης σύμφωνα με το αστικό δίκαιο. Και όλο και περισσότεροι άνθρωποι στην Πολωνία απασχολούνται στα πλαίσια των συμβάσεων του αστικού δικαίου και όχι με συμβάσεις δυνάμει του εργασιακού κώδικα. Ακόμα και ο εργασιακός κώδικας τα παγορεύει, αν κάποιος προσλαμβάνεται με μια σύμβαση δυνάμει του αστικού δικαίου, χρησιμοποιείται λοιπόν τα διαδικασία. Και ε, είναι απόλυτα νόμιμα αυτά, αυτές οι υποσχετικές. Τώρα, έχει αρμοδιότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γίνεται ανάθεση εξουσιών κανονικά. Πρέπει να υπάρχει ρητή αρμοδιότητα που δίδεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να κινηθεί. Όσον αφορά αυτό που συζητάμε, την προστασία των εργαζομένων, στην περίπτωση συγκεκριμένη, όταν λήξει η σύμβαση εργασίας, διότι εκεί χρησιμοποιούνται αυτές οι υποσχετικέ. Έχει αρμοδιότητα συγκεκριμένη Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα το άρθρο 153 των συνθήκων. Συμπληρωματική αρμοδιότητα, υποστηρικτική. Παρ' όλα αυτά, το άρθρο 153, παράγραφος 2, ρητά, δίνει την άδεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση να εκδίδει οδηγίε με ελάχιστες προϋποθέσεις για σταδιακή εφαρμογή αυτών. Προφανώ βεβαίω βεβαίω. και είναι τυπικό αυτό για τον τομέα αυτό, των συμπροματικών αρμοδιοτήτων μπορεί να εκδώσει και σύσταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχει αρμοδιότητα στον τομέα Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμω, κάτι πρέπει να υπογραμμιστεί. Όμω, σε αυτόν το τομέα είναι η ειδική νομοθετική διαδικασία που προβλέπεται. Χρειάζεται ομοφωνία. Και το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο απλώ εκφράζουν γνώμη. Όμω υπάρχει και ρήτρα πασαρέλα στη συνθήκη που επιτρέπει να περάσουμε στην κανονική νομοθετική διαδικασία αν το Συμβούλιο αποφασίσει ομοφόνο ούτω. Τελικά, πρέπει να θυμηθούμε ότι οι αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας σημαίνουν ότι για να κινηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να δικαιολογείται αυτό. Τα κράτη-μέλη δεν μπορούν να επιλύσουν το θέμα σε επίπεδο κρατών μέλων και ότι η δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα είναι αποτελεσματικότερη και αποδικότερη. Και σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, τα μέτρα που θα υθετηθούν δεν θα ξεπερνούν τα αναγκαία για την επίτευξη των καθοριστών των στόχων του άρθρου 153 να προσθέσουμε και κάτι. Ότι στη Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, και εδώ παίζει ρόλο αυτό, διότι αυτή η πρακτική της χρήσης αυτών των υποσχετικών, των λευκών, εναντίον των εργαζομένων μπορεί να θεωρηθεί ως παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, παραβίαση αξιοπρεπίας τους ή του δικαιώματος υπεράσπισής τους, διότι ο εργαζόμενος βρίσκεται σε μειονεκτική θέση σύμφωνα με την ομολογία του αστικού δικαίου. Η χάρτα απευθύνεται και στα κράτη-μέλη και στα θεσμικά όργανα την εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου. Αν θεσμικά όργανα αποφασίσουν, θετήσουν ε, όμω μια πράξη σχετική με αυτό το θέμα υπό τη μορφή οδηγία, τότε βέβαια αυτό θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα δικαιώματα που αγιώνονται στη χάρτα. Τέλο. Στο επόμενο τρίλεπτο ο Κροθυγό θα παρουσιάσω τη συγκριτική μελέτη την οποία συντόνισα στην ε, υπηρεσία έρευνα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με συμμετοχή αναλυτών πολιτικής από 11 χώρες. Ανέλησαν τις χώρες τους. Να δουν αν διαπίστωσαν παρόμοια προβλήματα στις χώρες τους όπως την Πολωνία. Καλύψαμε κάποιες δυτικοευρωπαϊκές χώρες, παλιά κράτη, μέλη, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ολλανδία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και κάποιες άλλες χώρες από την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, Ουγγαρία, Κροατία, Λετωνία, Λιθουανία και Ρουμανία. Και τώρα, όσον αφορά τις δυτικοευρωπαϊκές χώρες, τις παλιές ευρωπαϊκές χώρες, καταρχήν φαίνεται το πρόβλημα δεν υφίσταται εκεί. Ο ερευνητή που εξέτασε τη Γαλλία ανακάλυψε ότι δικαστήρια πάντα βλέπουν ένα ασφάλιο εργαζόμενο και σε κάποιε χώρε δεν είναι γνωστό, δεν υπάρχει νομολογία για την χρήση αυτό, των αξιογράφων. Η μόνη χώρα που ίσω να έχει παγκόσμιο προ πρόβλημα είναι το Ηνωμένο Βασίλειο. Διότι υπό κάποιου όρου το Βρετανικό Δίκαιο επιτρέπει στου εργοδότε να συμφωνήσουν να ζητήσουν την αποζημίωση και ίσω θα πρέπει ο εργαζόμενο να καταβάλει και το, την αμοιβή του για μια περίοδο. είχαμε την Cleveland ε, έναντι ε, Bluer με έναν μετανάστη Πολωνό που είχε υπογράψει ε, μια σύμβαση και αν εγκατέλειψε τη θέση του πριν από το προβλεπόμενο, έχανε όλες τις, όλους τους μισθούς. Το άτομο αυτό εργάστηκε κάποιους μήνες και μετά εγκατέλειψε πριν ολοκληρωθεί το χρονοδιάγραμμα και του στέρισαν τον ανθρώπου αυτού ε, τις αμοιβέ του. Η κυρία Μπρούερ πήγε στο δικαστήριο και έχασε στο, στο δικαστήριο γιατί έτσι προβλέπει το Βρετανικό δίκαιο, το Αγγλικό δίκαιο, από ό,τι φαίνεται. Τώρα, όσον αφορά τις χώρες Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, Στη Βουλγαρία ανακαλύφθη ότι η πρακτική που είναι γνωστή στην Πολωνία είναι γνωστή και στη Βουλγαρία. Υπάρχει νομολογία σχετική όπου αυτές οι συναλλαγματικές οι λευκές χρησιμοποιούνται στι εμπορικές, στις εργασιακές σχέσεις και υπήρχαν και κάποιες περιπτώσεις όπου ο εργοδότης ε, κέρδισε τη δίκη και έχασε ο Αυτή η κατάσταση συμβαίνει στη Βουλγαρία και παρόμοια πρακτική ακολουθείται σε Λιθουανία και Λετωνία. Κυρίως η Λιθουανία χρειάζεται περαιτέρω έρευνα, διότι υπάρχει δυνατότητα υπογραφή συμβάσεως με πλήρη ευθύνη, όπως ανακάλυψε ο ερευνητή που το βάρος της απόδειξης το μετακινεί. Μέχρι κάποιο ποσό θα πρέπει ο εργαζόμενος να αποδείξει ότι δεν έκλεψε τα χρήματα ή δεν κατέστρεψε εξοπλισμό. Επίσης στη Λετωνία ε, η ερεύνα απεκάλυψε ότι υπάρχουν συμφωνίες για υλικέ ευθύνε σύμφωνα με το δίκαιο, κάτι που υπογράφεται ξεχωριστά από ότι υπογράφεται στα πλαίσια του αστικού δικαίου, αλλά φαίνεται ότι δεν αποφασίζουν, είναι αποφάσει στον δικαστήρια. Κατακλείδη, το θέμα δεν ρυθμίζεται μέχρι τώρα από Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Προφανώ, όπω λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν υπάρχει καμία βάση η διαδικασία κατά παράβαση. Όμω, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αρμοδιότητα να δράσει στον τομέα σύμφωνα με το άρθρο 153 και θα μπορούσε να εκδώσει οδηγία και αυτή η πρακτική συμβαίνει σε πάνω από ένα κράτο μέλο όχι μόνο στην Πολωνία, αλλά στη Βουλγαρία και σε κάποιε από τι βαλτικέ χώρε. Αυτά και ευχαριστώ την προσοχή σα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μπάνκο. Ήταν σφαιρική, πολύ πλήρη η παρουσίασή σα από πλευρά ε, τη Επιτροπή και από τη Διεύθυνση Απασχόληση. Εγώ με την κυρία Μουριέλ ε, έχετε το λόγο για ένα πεντάλεπτο. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα πρώτα θα ήθελα να ευχαριστήσω ε, τους ετούντες την αναφορά, τους αναφέροντες τέλο πάντων γιατί πέσαν την προσοχή μας ε, σε αυτό το πρόβλημα. Ευχαριστούμε και το Κοινοβούλιο ε, για αυτές τις ε, αναλύσεις για την, τη συγκριτική μελέτη. Δεν θα σταθώ τώρα στα χαρακτηριστικά αυτής της συναλλαγματικής. Και αυτό το οποίο έχουμε λάβει υπόψη είναι ότι σε κάποιες περιπτώσεις ε, ε, βάσει της καλόπιστης συνεννόησης μπορεί να γίνει δαμόκλειος σπάθη αυτό το αξιόγραφο όσον αφορά τους εργαζομένους. Εφτά πολλές φορές γίνεται στο τέλος της σύμβασης εργασίας, οπότε αυτοί μπορεί να έχουν πρόβλημα και να μην μπορούν να αξιώσουν ε, το να απολάβουν των δικαιωμάτων τους ή καμιά φορά μπορεί να πολιτιστούν και από το να πάρουν τη σύνταξη. Οπότε ακριβώς όπως ε, αναφέρατε δεν υπάρχει στο κινητικό δίκαιο κάποια ρύθμιση για το πρόβλημα αυτό. Ο επομένως εδώ πέρα πρόκειται για μια αυθεντική περίπτωση επικουρικότητας. επίσης, υπάρχει μια ατμόσφαιρα απαγόρευσης για αυτήν την πρακτική στην Πολωνία ε, με χαρακτηριστικά πολύ συγκεκριμένα. Για μας είναι θέμα ε, υλοποίησης, εφαρμογής αυτών των κανόνων από τις ε, πολωνικές εθνικές αρχές. Δηλαδή, να μπορούν με επιθεωρήσεις, με, με τα δικαστήρια να εφαρμόσει να εφαρμόσουν οι Πολωνοί τέλο πάντων αυτό το οποίο προβλέπεται. Ούτω ώστε να διορθωθούν τα κακώ κείμενα. Είναι επομένως αυτό αρμοδιότητα των εθνικών αρχών. Όπως αναφέραμε και προηγουμένως δεν δικαιούται να πάνε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ούτε έχω σήμερα εντολή να σας πω σχετικά με την κοινοτική αρμοδιότητα. Θα πρέπει για να ε, συζητήσουμε για την νομική βάση να δούμε ακριβώς τι γίνεται με αυτό το έγγραφο το οποίο λάβαμε πρόσφατα. Γιατί θεωρητικά, όπως είδατε, μπορεί να έχουμε περισσότερες από μία νομικές βάσεις. Πάνω σε αυτό δεν μπορώ να σας σχολιάσω. Θα πρέπει πρώτα πρώτα να δούμε ποιος είναι ο σκοπός της ε, ρύθμισης. Καταλαβαίνουμε βέβαια ότι πρόκειται για πρακτικές οι οποίες δημιουργούν ε, σε διάφορα φυσικά πρόσωπα σημαντικές ε, ζημίες. Σας ευχαριστούμε κυρία Λέη Πρόεδρος και τώρα να δώσουμε το λόγο στους παρόντες Βουλευτέ. Η κυρία Πιτέρα, το λόγο. Με την ησυχία σας. Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Κοιτάξτε, εδώ κρύβεται το θέμα. Είναι και νόμιμο, είναι και παράνομο πρακτική αυτό. Η απόφαση του αυτοδικαστηρίου αναφέρει με σαφήνεια ότι δεν πρόκειται για νόμιμη πρακτική, αλλά δεν πρόκειται για δεσμευτικό δίκαιο, δεν δεσμεύει η δικαστική απόφαση. Γιατί για να αλλάξει πραγματικά η κατάσταση πρέπει να αλλάξει το αστικό δίκαιο. Να... Οι εργαζόμενοι στρέφονται προς τα δικαστήρια εργασιακού δικαίου. Και τελικά δεν έχουν οι επιστρέψεις εργασίας μέσα για να ελέγξουν το φαινόμενο αυτό ή για να επιβάλλουν κυρώσεις ενδεχομένω. Δεν υπάρχει απαγόρευση. Από την άλλη το φαινόμενο θεωρείται ότι δεν υπάρχει. Έγιναν κάποιε απόπειρε να απαγορευτεί αυτό το εργασιακό δίκαιο. Ξεκίνησε να επεξεργάζεται το θέμα το κοινοβουλίο μα. Δεν ολοκληρώθηκε όμω η διαδικασία αυτή. Και επειδή πρόκειται ακριβώς για ένα ευρύτατο φαινόμενο, Αφήστε που δε αυτή η μέθοδο εφαρμόζεται σε άτομα που δεν έχουν πάντα υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο, δεν έχουν απαραίτητα τι νομικέ γνώσει που χρειάζονται. Και γι' αυτό ανέφερε ο κ. ότι θα και αποφάσισε να υποβάλει ακριβώ την αναφορά και να στραφεί προ την Επιτροπή Αναφορών, γιατί γνωρίζει πολύ καλά ποια είναι τα προβλήματα που συνδέονται με το θέμα αυτό. Οι πιο πολλοί όμω ούτε τι γνώσει έχουν, τα χρήματα για να ζητήσουν την νομική σύνδρομη που χρειάζονται και δεν κατανοούν ότι αυτό αποτελεί μια παράνομη πρακτική. Υπάρχουν δικαστήρια που μπορούν να κοιτάξουν αυτά τα αξιόγραφα, τα γραμμάτια. Και συχνά τα ποσά είναι πολύ ψηλά. Και δεν υπάρχουν επαρκείς λοιπόν προδιαγραφές. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να καταθέσω επίσημα μια καταγγελία. Πρόκειται για μια ταπεινωτική και ευρέως δεδομένη πρακτική η οποία μειώνει τον εργαζόμενο και προτείνει λοιπόν την εξή λύση. Καταρχάς, και οι δύο σε αναφορές να μείνουν ανοιχτές. Κατά δεύτερον, να υπάρξει επαρκής πληροφόρηση η οποία να διαβιβαστεί και προς ε, την Επιτροπή μας. Κατά τρίτον, να αποσταλεί επιστολή προς την πολωνική κυβέρνηση και στο σχετικό Υπουργείο Εργασίας προκειμένου να τοποθετηθεί για το θέμα αυτό και με μια παράκληση να χορηγηθούν πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα τα οποία θα λάβει η πολωνική κυβέρνηση για να δοθεί ένα τέρμα στη διαδικασία αυτή, στο φαινόμενο αυτό. Και θα ήθελα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προετοιμάσει μια πρόταση ένα κανονισμό, μια οδηγία, μια απόφαση που θα σχετίζεται με το θέμα αυτό, που θα ασχολείται με το θέμα αυτό. Για ένα φαινόμενο το οποίο είναι διαδεδομένο ευρέως σε πρώην κομμουνιστικές χώρες και βλέπουμε λοιπόν ότι το παλιό σύστημα ε, εμφανίζεται ξανά και ξανά. Γι' αυτό λοιπόν ζητώ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, από τα νέα, από τα παλια κρατημέλη κράτη-μέλη, να μας βοηθήσουν να ξεφορτωθούμε επιτέλους αυτά τα παλιά υπολείμματα του κομμουνισμού. Και να δώσουμε και το λόγο στην κυρία Στανούκα. <clears throat> Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς να ευχαριστήσω <coughs> τους αναφέροντες που έθεσαν το θέμα. Καταρχάς Υποστηρίζω όλες τις δηλώσεις που έκανε ο συνάδελφος, μόνο ένα σχόλιο. Ο αστικός κώδικας, από ό,τι καταλαβαίνω, χρονολογείται το 1936. Η ίδια κατάσταση ισχύει και στη χώρα μου, στη Λετωνία, η οποία αναφέρθηκε στην έρευνα με την... θα γίνει μια αναβάθμιση μάλλον δεν έχει αλλάξει ο αστικός κώδικας από το 1937 μετά την εξαρτησία επανεφέρθη αυτός ο αστικός κώδικας. Και όλα τα μέσα και εργαλεία του δεν έχουν τροποποιηθεί και εμπεριέχουν αντιθέσεις όσον αφορά τη σύγχρονη νομοθεσία και την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως όσον αφορά τα δικαιώματα των εργαζομένων. Πρέπει να αποσταλεί επιστολή πράγματι στην Επιτροπή Απασχόλησης. Ήδη στον παρόδοτη με μέλος της. Είναι σημαντικότατο για μας να εξετάσουμε την κατάσταση και λυπούμε που περιοριστήκατε μόνο στην Πολωνία. Είναι σημαντικότατο να αποσταλεί η επιστολή προς τις πολωνικές αρχές. Πρέπει όμως να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά αυτή και να προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ κύριε Σανούκα. Κύριε Βαλέσα, θέλετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Υποστηρίζω πλήρως τα υποθέντα. Ακούσαμε μια τέλεια παρουσίαση. Δεν είναι μόνο πολωνικό πρόβλημα, αλλά όλου του ανατολικού μπλοκ των πρώην Σοβιετικών χωρών, των δορυφόρων της Σοβιετικής Ένωσης. Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε σαν παράδειγμα την Πολωνία, μεν είναι, δεν είναι γενικότερο πρόβλημα δε. Τούτου λεχθέντος υποστηρίζω πλήρως αυτά που είπε η κυρία Πιτέρα. Αυτά τα τρία βήματα δικαιολογούνται απολύτως. Να στείλουμε επιστολές στις ΔΕΟΣ στις αρμόδιες επιτροπές και να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προετοιμάσει περαιτέρω ανάλυση διότι είναι ε, υπάρχει παράδοξο. Κάτι είναι νόμιμα και παράνομο ταυτόχρονα. Ε, υπάρχει μια γκρίζα ζώνη στο νομικό τομέα. Δεν μπορούμε να τα αφήσουμε ως έχουν τα πράγματα και θα πρέπει σίγουρα να προχωρήσουμε στο θέμα αυτό. Ούτως ώστε να βγάλουμε μια άκρη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Μπελούστη, θέλετε το λόγο. Εσείς θέλετε το λόγο για Δύο λεπτά. E, Κυρίε και κύριοι, νομίζω ότι ουσιαστικά υπόθηκαν όλα τα απαραίτητα στοιχεία. Θα σας παρακαλούσα όμως να αναλογιστείτε τι θα γίνει για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό και μάλιστα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα σε περίπτωση που γίνει κατάχρηση των γραμματείων αυτών από πλευρά των εργοδοτών. Αυτό οικονομικά μπορεί να βαρύνει σημαντικά έναν εργαζόμενο, να προκαλέσει μεγάλα προβλήματα για να διαθέσει τα μέσα αυτά. Αλλά δεν έχω κάτι παραπάνω να πω. Σα ευχαριστώ απλά. Eh, σας ευχαριστούμε μέσα τη επιτροπής που ήρθατε για αυτή σας την υπόθεση που είναι τόσο σημαντική. Ενημερωθήκαμε για μέσω της ε, υπηρεσίας Έρευνα και είναι ένα θέμα το οποίο αφορά χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως αυτό το οποίο θέλουμε είναι να έχουμε ανοιχτή την ε, αναφορά και θα διαβάζουμε στην Επιτροπή τα υλικά που έχουν τόσο ώστε να γίνει αργότερα κάποια ανάλυση. Τι είπατε, τι είπατε. Ναι, πρόκειται για μια ανάλυση, γνωμοδότηση, στα ισπανικά έτσι το λέμε. Και επομένως θα πρέπει να δούμε ότι υπάρχει εδώ πέρα ασυμβατότητα, αλλά υπάρχει και παραβίαση του δικαίου. Επομένω θα συνονιθούμε με το Υπουργείο Εργασία τη Πολωνία και θα τους ε, πούμε ότι πρέπει να ξεκαθαρίσουν το γιατί έχει γίνει αυτή η κατάσταση, να μα πούνε τι θα κάνουν, πώ θα συνεχίσουν, με τι χρονοδιάγραμμα, τι διαβήματα θα αναλάβουν. Επομένως ε, θα κρατήσουμε την αναφορά ανοιχτή. Εντάξει, ωραία, συμφωνούμε πολύ. Ε, ευχαριστούμε κύριε Πελούς και τροπάμε στην επόμενη αναφορά προέρχεται από τον κύριο Κριστόμπαλ Αγουάδο Λάθα, Ισπανό. Εκπροσωπεί τον Γεωργικό Συνεταιρισμό της Βαλένθια Γεωργή Ασάχα και αφορά κάποια φυτογειονομικά προϊόντα. Βρίσκεται εδώ ο κύριος Λάθα. Έχετε πέντε λεπτά για να μας μιλήσετε για την αναφορά σας. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα σε όλους. Έξι αναφορές είχαμε υποβάλει σαν συνέχεια της ε, προβλημών της διαδικασίας για τις ε, ενεργές φυτογενομικές ουσίες. Οπότε και εμείς ε, θεωρούμε ότι δεν υπάρχουν τέτοιες εγκεκριμένες ουσίες ούτως ώστε να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε νόσους και οργανισμούς επιβλαβής δεν έχει δοθεί μια γενική λύση όσον αφορά ε, κάποιες καλλιέργειες οι οποίες δεν είναι πάρα πολύ κοινέ. Έτσι υπάρχει με κάποια γραμματεία στο Παρίσι, αλλά δεν χρηματοδοτεί τη σχετική έρευνα. Ούτε υπάρχει αμοιβαία αναγνώριση, γιατί σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα κράτη-μέλη δεν ενεργούν σύμφωνα με τον σχετικό κανονισμό. Επομένως, δεν υπάρχει συντονισμός και την πληρώνουμε εμείς οι γεωργοί. Αυτό το οποίο γίνεται ότι ε, ακριβώς ευλήξει συνέχεια ε, για την ίδια νόσο χρησιμοποιούμε το ίδιο φάρμακο υπάρχει αντίσταση του βλαπτικού οργανισμού. Έχει αποκτήσει ανθεκτικότητα. Είναι θέμα ποσότητας. Δεν, είναι πια θέμα ε, κάποιας περίπτωσης εξαιρετικής. Επομένως θα πρέπει να απαγορευτούν κάποιες αυτές τι ενεργές ουσίες. Αυτές που σήμερα επιτρέπουν να χρησιμοποιηθούν γιατί τελικά θα, δεν θα, έχουμε, ακόμα λιγότερα φάρμακα, λιγότερες συνδικές ουσίες. Θα πρέπει αυτό να το αντιμετωπίσει η Επιτροπή και τα κράτη-μέλη. Γιατί θα ζημιωθούμε εμείς οι γεωργοί. Θα πρέπει να συνοηθούν βέβαια τα κράτη-μέλη με την Επιτροπή. Έχουμε και άλλη μία ε, θέση όσον αφορά τώρα την αύξηση αυτών των χωρών, ε, τη χρήση μάλλον αυτών των ουσιών από, από προϊόντα που εισέρχονται από τρίτες χώρε. Οπότε θα πρέπει να δούμε το πώ θα υπάρξει ένα ε, καινούριο κανονισμός κανονισμό και να είναι πιο αυστηρός όσον αφορά του σχετικού ελέγχου για τα προϊόντα που έρχονται από τι τρίτε χώρε. Ελπίζουμε αυτό να γίνει και να έχουμε έναν κανονισμό πιο ρεαλιστικό, αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει τις κατάλληλες αποφάσεις, ούτω ώστε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Να μην κάνει ό,τι τα τελευταία χρόνια. Γιατί εκτός από τα κενά του ισχύοντος κανονισμού, δεν έχουμε την φυτογενομική ασφάλεια που απαιτείται. Δεν ήταν η αποφασιστική επιτροπή ανάλογα με την ε, σημασία και υπάρχει αυτή η αρρώστια του, της μαύρης κοιλίδας στα εσπεριδοειδή. Υπήρξε μεγάλο πρόβλημα. Είχαμε από την Νότιο Αφρική 16 κρούσματα, 16 από την Αργεντινή και 70 από τις αγωγές από την Ουρουγουάη. Και αυτά είναι στοιχεία της ίδιας Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και επομένως ε, αυτή η χαλαρότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μας έφεραν στο χείλος του γκρεμού. Οπότε είδαμε τώρα σε πόσο πόσο αυτό το πρόβλημα ε, μας οδήγησε σε εξάπλωση αυτών των ασθενειών ε, και μάλιστα των ασθενειών των χειρότερων σε όλο τον πλανήτη. Εξαπλώνει την Ευρωπαϊκή Ένωση, στη Βόρεια Ισπανία, στην Πορτογαλία υποφέρουμε μεταξύ 2013-2014 είχαμε 19 κρούσματα αυτής της ασθενείας. Πρόκειται για διάφορες ε, ασθένειες επίσης που αφορούν τα εσπεριδοειδή και 16 Δεκεμβρίου του 2014 ε, εξέδωσε ένα κείμενο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είπε ότι θα πρέπει να υπάρχουν κάποιε δαπάνε ούτω ώστε να καταπολεμηθούν αυτοί, αυτοί οι βλαβεροί οργανισμοί. Και είπε ότι το 2013 είχαμε τουλάχιστον οκτώ τέτοιες ασθένειες για τα φυτά. Και έτσι κάθε επτά μήνες είναι σαν να έχουμε ε, μια καινούργια επιθυμία. Το θέμα είναι αν η τελική απόφαση θα ληφθεί επί τη βάση μιας μελέτης του κινδύνου από την ε, ΕΦΣΑ, ε, την Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων ή από την Μόνια Επιτροπή. Και έχουμε τώρα μια τρίτη αναφορά, το πώς θα πάρουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, δεν θα έχουμε ανοχή των όσων εισάγονται από τις τρίτες χώρες γιατί γνωρίζουμε ότι από πλευράς εμπορικής δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχουν αυτού του είδους τα περιθώρια ανοχής της εισαγωγή, γιατί τότε θα υπήρχε μεγάλη ζημία των κρατών μελών οπότε θα πρέπει να υπάρχει κάποια αμοιβιότητα. θα έπρεπε πάντως λόγω της αμοιβιότητας ακριβώς ό,τι απαιτείται από τους ε, Ευρωπαίους γεωργούς τις ίδιες ε, απαιτήσεις να τις έχουμε και για τους γεωργούς που μας εξάγουν το πρόγραμμα. τους. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε. Τώρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μας πει σε σχέση με αυτήν την αναφορά. Πρώτα η κυρία Πιτών. Στη συνέχεια θα λάβει το λόγο ο κύριος Γιάννης Καραμίσιος. Έχετε Πέντε λεπτά ο καθένα για να μα ενημερώσετε. Yes, thank you. Σας ευχαριστώ. πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο. Καταρχάς θα ήθελα να απαντήσω στα θέματα που τίθενται στην πρώτη αναφορά. Αυτό το έχουμε άλλωστε εξετάσει και στο παρελθόν και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δώσει και ενημερωτικά στοιχεία σε ό,τι αφορά την ε, ε, την απόσταση της νομοθεσίας αυτής που έχει να κάνει με το θέμα αυτό. Και σήμερα λοιπόν βρισκόμαστε σε ένα εντελώς καινούριο ε, νομοθετικό πλαίσιο με τον κανονισμό 2009, ο οποίος ε, εφαρμόστηκε καθ' ολοκληρία τον Ιούνιο του 2011 και πιστεύουμε ότι είναι σαφής σε σχέση σε ό,τι αφορά τις προθεσμίες για τη διαδικασία, για την έγκριση ενδεχομένως των δραστικών ουσιών και για τα θέματα αυτά της διαδικασίας. Ως εκ τούτου, το πρόβλημα που αναγνωρίζουμε και το οποίο υπογραμμίζει ο ετών σε ό,τι αφορά την καθυστέρηση και την εφαρμογή της αμοιβαία αναγνώρισης από τα κράτη-μέλη, παρακολουθείται και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή χάρη στο έργο των συναδέλφων της τις Υπηρεσίας και πραγματικά παρακολουθούμε την κατάσταση για να βρούμε μια λύση και για να παρατρύνουμε τα κρατημέλη να σεβαστούν τις προθεσμίες και τις διατάξεις του κανονισμού σε ό,τι αφορά τις ίσονος σημασίας χρήσης. Χαίρομαι που ο συντονιστικό οργανισμό ξεκίνησε να εργάζεται το Σεπτέμβριο του 2015. Αναμένουμε μια διάμεση αναφορά συντόμω. Αυτή λοιπόν η υπηρεσία συντονισμού αναζητά τι λύσει, ε, τι τεχνικέ, ε, χημικέ και μη για τα κράτη-μέλη για την αντιμετώπιση ε, των ζυζανίων ε, στις μικρές καλλιέργειες προκειμένου και η διαδικασία εγκρίσης και ε, είναι σε συνδυασμό με το IPM που περιλαμβάνει διάφορα έργα και αυτό λοιπόν ε, θα δώσει απάντηση στα πιο πολλά ζητήματα που συνδέονται με τις μικρές καλλιέργειες, με τους μικρούς καρπούς. Ελπίζουμε λοιπόν ε, σύντομα να βρούμε μια σχετική λύση για το θέμα αυτό. Σε ό,τι αφορά λοιπόν το θέμα αυτό, θα ήθελα να, ενημερώσω τον αναφέροντα ότι αναγνωρίζουμε ότι τα στοιχεία του κανονισμού μπορούν να, να επεκταθούν περαιτέρω και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην τρέχουσα φάση ε, και σε σχέση με τον κανονισμό 36 του 2005 είναι σε ε, φάση αξιολόγησης, refit και η αξιολόγηση των δύο νομοθετημάτων θα γίνει στο εγγύς μέλλον. Και η δημόσια διαβούλευση αναμένεται ότι θα ξεκινήσει ήδη μέχρι το τέλος του χρόνου. Σε ό,τι αφορά τα περαιτέρω στοιχεία, το τρίτο τμήμα της ε, αναφοράς, σε ό,τι αφορά την ανοχή εισαγωγής, να ενημερώσουμε την Επιτροπή ότι πρόκειται για μία αρχή βασική για το διεθνές εμπόριο, αυτή η αρχή της ανοχής εισαγωγής. Και πιστεύουμε λοιπόν ότι θα πρέπει να εφαρμόζεται πλήρω από την Ευρώπη και από τις χώρες που εισάγουν στην Ευρώπη. Πρόκειται για καρπούς που δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση. Συνδέεται όμως με την ε, ασφάλεια του καταναλωτή και ε, περιοριζόμαστε μόνο τις περιπτώσεις όπου αποδεικνύεται η ασφάλεια της χρήσης. Ε, θα προεριστώ λοιπόν στα στοιχεία αυτά και θα δώσω το λόγο στον συνάδελφο για το δεύτερο τμήμα της αναφοράς. With uh, respect... Όσον αφορά το θέμα των μαύρων κελίδων στα σπεριδοειδή, έχουμε ανησυχητική τάση. Είδαμε πολλές περιπτώσεις στην Αργεντινή, στην Ουρουγουάη, την Νότια Αφρική. Βρήκαμε αυτό το παράστο. Θα λάβει μέτρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά την Αργεντινή και την Ουρουγουάη. Η μόνιμη διαρκή Επιτροπή το ζητά αυτό και επιθεωρητέ τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα επισκεφτούν τι εν λόγω χώρε σύντομα για να εξετάσουν επιτόπου ποια είναι η κατάσταση. Όσον αφορά το πρασίνισμα των εσπεριδοειδών, έχουμε την αυστηρότερη προσέγγιση στην νομοθεσία μα είναι ένα παράσιτο το οποίο δεν επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει καραντίνα. Τα εσπεριδοειδή που καλλιεργούνται εκεί που υπάρχει το παράσιτο δεν εισάγονται. Ούτε εσπεριδοειδή με φύλλα που μπορεί να έχουν αυτό το παράσιτο πάνω τους. Και φορέας του παρασίτου αν έχει την καλωσία μου δώστε λίγο χρόνο να εξηγήσω Ξέρουμε ότι φορέας του παρασίτου αυτού βρίσκεται στη Γαλλικία της Ισπανίας και στην Πορτογαλία. Από ό,τι ξέρουμε δεν έχουμε όμως μια επιδημία, δεν έχει εμφανιστεί κρούσμα με πολλά παράστα στην Ευρώπη. Έχουν λάβει επίγοντα μέτρα στην Πορτογαλία και θα παρακολουθήσουμε σαν Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι γίνεται, πώς εφαρμόζονται τα μέτρα εκτάκτου ανάγκης. Και αν υπάρχει κάποιο ξέσπασμα της και ο κίνδυνος αυξηθεί, θα ληφθούν τα ενδεδειγμένα μέτρα. Για την ώρα όμως, και το επαναλαμβάνω από ό,τι γνωρίζουμε, δεν έχουμε ε, ένα ξέσπασμα, μια επιδημία. Βασιζόμαστε στα κατεπήγοντα μέτρα ε, τα οποία έχουν κοινοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τέλος, γενικότερα, ένας νέος κανονισμός για τα φυτογενομικά εγκρίθηκε σε πολιτικό επίπεδο από Κοινοβούλιο και Συμβούλιο. Ο τελευταίος τριμερής διάλογος έλαβε χώρα το Δεκέμβριο. Το κείμενο θα ετοιμαστεί, σύντομα θα παρουσιαστεί στην Επιτροπή Γεωργίας ε, για ψηφοφορία. Στο κείμενο θα δείτε ότι έχουν ενισχυθεί οι κανόνες περί εισαγωγών. Και ένας από τους κανόνες αυστηρότερους είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να θετήσει εντός διετίας από τη θέση σε ισχύ των λόγω κανονισμού κατάλογο φυτών υψηλού κινδύνου που θα απαγορεύεται η εισαγωγή τους βάσει μιας προκαταρτικής αξιολόγησης μέχρι ότου αποδειχθούν ασφαλή. Υπάρχουν και άλλα αυστηρά μέτρα που θεσπίζονται όπως απέτηση για υγειονομικό πιστοποιητικό για την εισαγωγή όλων των φυτών, καρπών και λαχανικών, φρούτων και λαχανικών, ένα νέο σύστημα που πιστεύουμε ότι θα κάνει πιο αυστηρού κανόνες εισαγωγής και θα προστατεύσει την Ευρωπαϊκή Ένωση έναντι εισαγωγών, παρασίτων και ενώσεων από τρίτες χώρες. Ευχαριστώ κύριε Καραμίτσο. Και τώρα, οι συνάδελφοι που έχουν ζητήσει το λόγο. Κύριε Αλμπιόλ, πρώτη σα ευχαριστώ πολύ, λέει κυρία Αλμπιόλ. Πρώτα-πρώτα να ευχαριστήσουμε του αναφέροντε που ε, υπέβαλαν την ε, αναφορά στην Επιτροπή μα. Θα πρέπει να σα πω δύο την όσον αφορά τα θέματα τα οποία έθεσαν οι αναφέροντες ε, όσον αφορά τον ε, έλεγχο για τις αρρώστιες. Αυτό είναι ένα σωστό βήμα ε, και θα πρέπει να είμαστε πιο αποτελεσματικοί οπότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να λάβει τις κατάλληλες αποφάσεις και ούτως ώστε να αρθούν τα κενά του ισχύοντος κανονισμού. Νομίζω, όπως ακριβώς είπαν οι αναφέροντες, ότι Έχουμε τώρα έναν κανονισμό και κάποιες πολιτικές αποφάσεις ε, που οδήγησαν στο να έχουμε τις συγκεκριμένες ασθένειες που έχουν εισαχθεί στην Ευρώπη και οι οποίες έχουν ε, επεκταθεί όπως είπαν οι αναφέροντες αλλά θα πρέπει να αφήσουμε ανοιχτή την αναφορά και θα πρέπει να δούμε το πώς θα λειτουργήσει ο νέος κανονισμός και να αξιολογηθεί κατά πόσον αυτός ο ε, κανονισμός αποδίδει δεν αποδίδει. Ας μείνει ανοιχτή η αναφορά. Και επίσης νομίζω ότι το σωστό είναι να ζητηθεί ότι τα εισαγόμενα προϊόντα ε, θα υπάγονται στις ε, ίδιες προϋποθέσεις όπως και τα δικά μας ε, προϊόντα τα οποία παρέχουν περισσότερες εγγύησεις. Οπότε έτσι νομίζω ότι θα καταλήξουμε σε αυτά τα οποία ζητούν οι αναφέροντες. Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη ο προβληματισμός για το τι θα γίνει, θα πρέπει να γίνει η αξιολόγηση του νεοκανονισμού και των νέων μέτρων και ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε κυρία Αλμπιόλ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστούμε τους ε, αναφέροντες και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα συμφωνεί με τα όσα ζητήσαν και είπαν κατά κάποιο τρόπο ήταν απογοητευτικά όσα είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, δεν δώσαν λύσεις σε τρία βασικά σημεία τα οποία υπάρχουν και είναι παλαιά αιτήματα αυτά. Πρώτα πρώτα είπαμε για την σπάνη των ενεργών ουσιών. Όλοι γνωρίζουμε ότι έχει μειωθεί ο αριθμός των ενεργών ουσιών. Και επίσης έχουμε οδηγηθεί σε αύξηση της ανθεκτικότητας των ε, ιών, των ασθενειών τέλο πάντων. Δεν κάνει τίποτα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχει κάποιες ειδικέ διαδικασίες που οδήγησαν σε αυτά τα αποτελέσματα. Άρα θα πρέπει να, ε, να αναρωτηθούμε τι γίνεται για αυτό το πρόβλημα. Άρα θα πρέπει να βρεθεί σύντομα λύση. Οπότε αυτό θα ρωτήσω εγώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τι κάνει, τι κάνει γι' αυτό, τι θα γίνει στο μέλλον. Έχουμε τώρα αυτό το καινούριο ταμείο του που συγκροτήθηκε τον ε, Σεπτέμβριο του 2015. Είπαμε ότι θα πρέπει να δούμε αν μπορούμε να έχουμε αδειοδότηση για νέες ενεργές ουσίες και αυτές να είναι χρήσιμες. Τώρα για να δούμε τι γίνεται όσον αφορά τα εφαρμοζόμενα, τα χρησιμοποιούμενα κατάλοιπα και τις ουρακές τιμές. Θα πρέπει να υπάρχει αμοιβαιότητα σε σχέση με όλα αυτά, σε σχέση με τις εισαγωγές. Αυτά τα οποία ζητεί η Ευρωπαϊκή Ένωση από τους ε, δικούς μας παραγωγούς να τα ζητά και από τους παραγωγούς των τρίτων χωρών. Ε, επίσης σας λέω ότι με απασχολεί αυτό το οποίο απάντησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι τόσο σοβαρό το θέμα που απαιτεί αποφασιστικότητα. Θα πρέπει να γίνει εξολόγηση των κανονισμών. Θα πρέπει να γίνει δημόσια διαβούλευση κατά τα τέλη του έτους. Αλλιώς θα συνεχίσουμε τον ίδιο τρόπο. Θα συνεχίσουμε τα ίδια προβλήματα. Θα συνεχίσουμε να εισάγουμε χωρίς νομοθεσία, χωρίς ε, ελέγχους τα προϊόντα από τρίτες χώρες. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να ενεργήσουμε άμεσα και να ληφθούν μέτρα ε, και για τα κατάλοιπα και για τα υπόλοιπα προβλήματα πριν τα τέλη του έτους. Άρα νομίζω ότι θα πρέπει να μας εξηγηθεί σε αυτήν την καινούρια μαύρη λίστα τι γίνεται, ποιοι είναι οι κίνδυνοι. Είδατε το πρόβλημα με την μαύρη χιλίδα. Είναι πολύ επικίνδυνη ασθένεια. Είπαμε ότι ε, ακόμα δεν είχε έρθει. Αλλά τώρα ο κίνδυνος είναι μεγάλος να εισαχθεί. Και αυτό να το μετανιώσουμε πικρά στην συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μάτο, λέει η Πρόεδρος. Δεν ξέρω εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει κάτι να διευκρινίσει κάτι το οποίο θα μπορούσε να φωτίσει περισσότερο αυτές τις ε, ε, αμφιβολίες που υπάρχουν. Θέλει κάποιος να διευκρινίσει, έχετε το λόγο. Thank you, Madam Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Για ένα λεπτό να διευκρινίσω το θέμα του νέου κανονισμού για τα μέτρα κατά των ε, παρασύτων των φυτών. Έγινε διαβούλευση πριν υποβάλει πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή του κανονισμού συζητήθηκε εκτενώς από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κανονισμός και συμφωνήθηκε ότι το εισαγωγικό καθεστώς πρέπει να παραμένει, να διαμορφώνεται βάσει του κινδύνου. Θα είμαστε αναλογικοί, θα επικεντρωνόμεθα επί των κινδύνων και θα είμαστε και δραστήριοι, ενεργοί. Δεν είναι δυνατόν, δεν είναι, δεν είναι δεκτόν από τι εμπλεκόμενους φορείς να αποκλείσουν τις εισαγωγές εντελώς. Δεν θα είναι ανάλογο προς τον κίνδυνο που αντιπροσωπεύουν ε, πολλά φρούτα και φυτά που εισάγονται. Αν δούμε προβλήματα όπως στην περίπτωση Αργεντινής και της Ουρουγουάης ή όταν διαπιστώνουμε προβλήματα όσον αφορά λαχανικά που έρχονται από την Ασία, όπως κάναμε και σε πολλές άλλες περιπτώσεις, μπορούμε να λάβουμε τα ενδεδειγμένα μέτρα και σε κάποιες περιπτώσεις μπορούμε να απαγορεύσουν εισαγωγή φυτών αν βάση αξιολογήσεως κινδύνων αποδεικνύεται ότι δημιουργούν απαράδεκτο φυτογενομικό κίνδυνο για την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ κύριε Καραμίτσιο για να ολοκληρώσουμε. Κύριε Αγουάδο, για να ολοκληρώσετε από πλευρά των αναφερόντων. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρώτα πρώτα. Συνεχίζει και δεν βρίσκει λύση σε σχέση με την αμοιβιότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να δούμε αν θα λυθεί το πρόβλημα στο μέλλον. Αλλά όμω τόσα χρόνια λέμε τα ίδια. Ενώ το είπαν πρόσωπα που τα σέβομαι πάρα πολύ. Όμω για το δεύτερο σημείο θα ληφθεί κάποια απόφαση με επιστημονικά ή με πολιτικά κριτήρια. Για μένα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μα απασχολεί πολύ αυτό. Για το τρίτο σημείο τώρα, ουδέμια λύση προτείνεται. Δηλαδή τι γίνεται σε σχέση με τον αθέμητο ανταγωνισμό που υφιστάμεθα οι Ευρωπαίοι. Όταν εμείς εξάγουμε σε τρίτες χώρες, Φερρυπίνης της ε, είπα μας απαιτείται, ε, απαιτούν από εμάς μάλλον να υπαχθούμε στις ε, προϋποθέσεις που εκείνοι τάσουν. Αυτό μας ενοχλεί πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Βάδο. Ήρθε ο κύριος Ζόρντι Σεβαστιάν, ο οποίος νομίζω ότι θέλει να μιλήσει και αυτός. Έχετε ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε συμπαθάτε με που καθυστέρησα. Αλλά έχει, δεν είναι σημείο στη σωστή ώρα. Ελπίζω να κρατήσουμε ανοιχτή αυτή την αναφορά. Κυρίως και που δεν άκουσα τη συζήτηση. Όσον αφορά επομένω αυτές τις ενεργές ουσίες, όταν ορίζει ε, κάποιο είδου εξαιρετική ε, ρύθμιση ο, ο κανονισμός και όταν όμως συνεχίζουμε να έχουμε το πρόβλημα, αυτό σημαίνει ότι ο κανονισμός δεν αποδίδει. Κατ' εξαίρεση η ρύθμιση σημαίνει όταν κάτι γίνεται ε, αραιά και πού, όχι όμως συνέχεια. Τώρα όσον αφορά αυτά τα μέτρα όπως τα μέτρα της αμοιβιότητας, το θέμα είναι εάν υπάρχει δημοσιονομική υποστήριξη για να γίνει έρευνα και να δούμε κατά πόσο η εξαιρετική χρήση των φαρμάκων ε, μπορεί να υποστηριχθεί. Σε κάποιες επαρχίες και περιφέρειες ο κόσμος εξαρτάται από την γεωργική παραγωγή απολύτως. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό το τι επιτρέπεται και τι δεν επιτρέπει πλευράς φυτοϊγειονομικής, φυτοπροστατευτικής. Έχουμε θέμα τον ανταγωνισμό. Εάν ε, πρέπει η δική μας ε, παραγωγή να εφαρμόσουν περισσότερα από όσο οι ανταγωνιστές. Δεν είμαστε ανταγωνιστικοί με αυτόν τον τρόπο. Θα πρέπει να, να είναι ο ανταγωνισμός τίμιος. Επίσης θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι αυτά τα μέτρα και την υγεία και το περιβάλλον. Κύριε Σεβαστιά, σας ευχαριστώ. Ως συμπέρασμα των όσων άκουσα εδώ. Νομίζω ότι συμφωνούμε. Θέλετε και εσείς το λόγο κύριε Σπάτα. Ναι, ναι, ναι, ναι. Ένα λεπτάκι γιατί πριν δεν το είπα. Είναι δεδομένο το εμπάρκο με τη Ρωσία, αλλά θέλω να συμφωνήσω με αυτά τα οποία είπε η συνάδελφος ε, Αλμπιόλ. Να μείνει ανοιχτή η αναφορά, αλλά να κάνουμε και κάτι παραπάνω, να απευθυνθούμε στην αρμόδια επιτροπή, να αναζητήσει λύσεις, να κάνει κάτι για αυτή την κατάσταση της σπάνιδος των ενεργών ουσιών. Επίσης να δούμε κατά πόσον ε, είναι δυνατόν να αναβαθμιστεί το ταμείο για το οποίο συζητούμε και επίσης θα πρέπει κάτι να γίνει όσον αφορά και τη, τις προϋποθέσεις υποκαθεστώς ε, αμοιβιότητας. Έλεγα, συμπεράσματα, υπάρχει σαφή συνένεση ότι αφού τώρα είναι ε, επικρέματα από την έγκληση του κανονισμού θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι μελετήθηκαν όλες οι δυνατές λύσεις αλλά εάν δεν έχετε αντίρρηση να διαβιβάσουμε το υλικό στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ξέρουμε πότε θα ολοκληρωθεί η δικασία του κανονισμού αλλά θα πρέπει να ενημερωθούμε Αυτά τα οποία λέει αναφορά θα τα καλύψει ο κανονισμός, θα τα καλύψει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με τι χρονοδιάγραμμα. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο πρόβλημα της γεωργίας και του περιβάλλοντος. Είναι πρόβλημα και ανταγωνισμού. Επομένω θα πρέπει να δούμε τι θα πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν της διαβάσουμε όλο αυτό το υλικό παρακαλούμε να μας απαντήσει με κάποια μικρή έκθεση για το πώς έχουν τα πράγματα αλλά και να απαντήσει και για τα θέματα ανταγωνισμού. Συμφωνείτε? Ευχαριστώ πολύ κύριε Αγουάδο. Θα είμαστε σε επαφή για να παρακολουθήσουμε την εξέλιξη της υπόθεσης. Καλώς. Λέει η πρόεδρος. Και τώρα. Τρίτη αναφορά τη σημερινή απογευματινή συνεδρίαση. Ε, αναφορά Άγχελ Ερνάντεθ Λορέντο, Ισπανία. Εκ μέρου του Συνδικάτου Κομισιόνε Ομπρέρα τη ε, Λεόν. Αφορά την δόλια εκαθάριση του εργοστασίου Πουέρτα Νόρμα στη Σόρια τη Ισπανία. Εδώ παρίσταται ο κύριο Ερνάντεθ Λορέντο. Καλώ ορίσατε. Έχετε ένα πεντάλεπτο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Καλησπέρα σα. Αυτή η αναφορά υπευλήθη το 2013 τον Μάρτιο. Αφορά αυτή την ε, πτώχευση αυτού του εργοστασίου. Ασχολείται με την κατασκευή ξύλινων πορτών ε, στην κοινότητα Σαν Λεωνάρδο Δεγιάγουε, στην ε, αυτόνομη διοικητική περιφέρεια Στήγια Ηλαιών. Ο, ο πληθυσμός ανέρχεται σε 2.300 κατοίκους και όλη αυτή η επαρχία έχει 23 κοινότητες και 15.000 κατοίκους και αυτή η δραστηριότητα, δηλαδή η εκμετάλλευση του δάσους και της ξυλίας είναι βασική ε, πηγή επιβίωσης αυτών των ανθρώπων. Το 1992 ε, αυτή η εταιρεία που δείχνει το 55 και είχε 800 εργαζομένους ε, πουλήθηκε στην εταιρεία στον Όμιλο Yeld Ven πάρα πολύ ε, μοντέρνα η πιο μοντέρνα λέγανε τέτοια εταιρεία στην Ευρώπη και είχε πάρει από την περιφερειακή κυβέρνηση επιδοτήσεις και επιδοτήσεις αυτές προέρχονται από το Ταμείο Περιφερειακής από το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και είπαμε ότι αυτή η εταιρεία το 2011 έκανε αίτηση ε, πτώχευσης. Το 2012 ξεκίνησε η εκαθάριση ε, της εταιρείας αυτής. Ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2013 και υπήρξε ε, δικαστική απόφαση όσον αφορά την εκποίηση των εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού γενικά και αυτό έγινε από τις αρμόδιες αρχές της Σόρια. Και ε, τώρα ε, αγοράστηκαν όλα αυτά από την Norma Doors Technologies και μια εταιρεία που έχει πάρα πολύ σημαντική ανάπτυξη οπότε εκεί έπιασαν 250 εργαζόμενοι και υπήρξε ανάλυση επομένως αυτή της, εταιρεία, της, ε, της, της αίτησης ε, πτώχευσης. Οπότε είπαμε ότι αυτή η εταιρεία ακολούθησε κάποια στρατηγική και γι' αυτό ήθελε να εκρήσει πτώχευση, να κάνει εκαθάριση στην θηγατρική και το ίδιο έκανε και σε άλλες επιχειρήσεις αυτής της ομάδας, αυτής της, ε, του ομίλου τεριών Και ε, όλοι αυτοί επομένω προχώρησαν σε πτώχευση και καθάριση Οπότε διάφοροι ευρωβουλευτές και ε, κάποιοι από την Επιτροπή κατάφεραν να γίνει κάποιο είδους συλλογική ε, συμφωνία ε, μεταξύ εργαζομένων ε, και, του ομίλου αυτού, Τζέλντ Βεν. Οπότε άμεσα και χωρίς καμία καθυστέρηση δόθηκαν οι αποζημιώσεις που έπρεπε σε αυτούς τους εργαζομένους μια που πια δεν είχαν σύμβαση εργασία. Οπότε αυτή η εταιρεία Τζελτ Βεν στα πλαίσια των κοινωνικών τους υποχρεώσεων δώσαν 500.000 σε κάποιο ίδρυμα στην ε, Λεόν και στην Καστία και Λεόν τέλο πάντων για να βοηθήσουν την επανεγκατάσταση των εργαζομένων. Και ε, βοήθησε γενικά η κοινότητα της Καστήλης και Λεόν με τη βοήθεια του Ευρωπαϊκού Ταμείου Παγκοσμιοποίησης και Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το, ποσό για το οποίο συνέβαλαν ανέχεται σε 700.000 ευρώ. Παρ' όλα αυτά, όταν ε, ε, επιλήθηκε αυτή η διαφορά, και ε, αυτή, αυτή η διαφορά έδειξε ότι υπάρχουν κάποια παραθυράκια στο κοινοτικό δίκαιο. Υπάρχουν κενά στο δίκαιο για, για τα προβλήματα των ε, επιχειρηματικών ομίλων. Υπάρχουν προβλήματα στην κάλυψη από τα ευρωπαϊκά ταμεία. Ε, και έτσι είναι, αυτό είναι κάτι το οποίο βλάπτει το βιομηχανικό ιστό. Θα πρέπει επομένω ο Ευρωπαίος νομοθέτης να βρει κάποιες λύσεις. Ο κανονισμός του 2015 υπαρχμόν 848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Μαΐου του 2015 ε, περιέχει κάποιες σχετικές διατάξεις, δηλαδή για κάποιες ε, εταιρείε που ανήκουν στον ίδιο όμιλο. Για, να, ε, περίπτωση που έχουμε δύο ή περισσότερες επιτοχεύσεις που είναι συναφείς οικονομικά και που προέρχονται όπως είπαμε από τον ίδιο όμιλο εταιριών. Είπαμε για κάποιες ε, παράλληλες διαδικασίες που θα πρέπει να περάσουν από τη διαδικασία και την αρχή της ε, ισότητος. Όμως, αυτός ο κανονισμός δεν καλύπτει κάποιες άλλες περιπτώσεις, γιατί πολλές φορές κάποιες ε, εταιρείε που κάνουν αυτή την πρακτική από νομικής πλευράς είναι άσχετες μεταξύ τους, αλλά συνδέονται από πλευρά και οικονομικέ. Και έχουμε επομένω μια εταιρεία που περνά από τη διαδικασία τη πτώχευση, ενώ οι άλλε ε, όχι. Οπότε αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι αυτή η νομοθεσία δεν περιέχει διατάξεις ούτω ώστε να αριθμίζονται ε, τέτοιες περιπτώσεις δόλιας πτώχευσης. Και πρέπει να γίνει ε, μια παράλληλη διαδικασία, μια συντονισμένη διαδικασία. Εμείς αυτό το οποίο λέμε και θεωρούμε ότι είναι προς το μας είναι να έχουμε ενιαίες διατάξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση διατάξεις που να προβλέπουν ακριβώς την ευθύνη ε, όλων των εταιριών ενός ομίλου εταιριών και έτσι ε, να ρυθμίζεται τι γίνεται με τα χρέη αυτών των εταιριών και ε, να, όταν έχουμε καθάριση κάποιας εταιρεία ή όταν έχουμε κάποια μετεγκατάσταση θα πρέπει να υπολογίζεται ε, το, το κόστος και να προβλέπεται διακόπτη ο, η πρόεδρος. Παρακαλώ ολοκληρώστε. Ναι, ναι, ναι λέει. Ε, έχουμε την υπόθεση Budget που εξετάζεται από την Επιτροπή ΟΣΑ και την ε, έκθεση Winter του 2002. Θα πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτά να τα λάβει υπόψη, να προβεί κάποια ρύθμιση, όπως και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε έναν νέο ε, κανονισμό για την κοινωνική επιχειρηματική ευθύνη. Και θα πρέπει όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία σα επισημάναμε να ληφθούν υπόψη και σα ευχαριστούμε. Εμεί ευχαριστούμε. όπω γνωρίζετε, έχει ζητηθεί η σχετική γνωμοδότηση από την Νομική Επιτροπή. Νομίζω δεν έχετε παραστήσει στην ε, συνεδρίαση την σχετική, οπότε θα πρέπει να σας διαβιβάσουμε ό,τι στοιχεία έχουμε. Γιατί ε, μελέτησαν το θέμα ε, τα μέλη της, Επιτρο... της νομικής επιτροπής, ο κύριος, αυτό που, όλα αυτά που είπε ο κύριος Ερνάντες του Συνδικάτου Κομισιόνες Ε, εμείς πρέπει να σας πούμε ότι είμαστε αλληλέγγυοι για τους 500 και πλέον ε, εργαζομένους οι οποίοι έχασαν τη δουλειά τους ακριβώς επειδή έκλεισε λόγω της πτώχευσης ε, το εργοστάσιο. Ξέρει η Επιτροπή μας το πόσο αρνητικά αποτελέσματα έφερε το κλείσιμο του εργοστασίου. Τι κακό ήταν αυτό για την ε, ευημερία της ε, περιοχής. Τι έγινε με όλους αυτούς που χάσαν τη δουλειά τους. Τι έγινε με... Πόσο αρνητικό ήταν αυτό για την περιοχή αυτή της Σόρια. Έχουμε τώρα αυτήν την πολυεθνική, αυτήν την μητρική εταιρεία του, του Πουέρτας Νόρμα. Ε, ήταν η εκαθάριση δόλια και η μητρική εταιρεία αυτό το οποίο ήθελε με τη δόλια καθάριση είναι να κλείσει το εργοστάσιο για να με την κατασταθεί η επιχείρηση. Ζητεί επομένως ε, ε, ζητεί ο, αναφέρον να αναγνωριστεί το ότι η μητρική εταιρεία παρέβει τον κανονισμό 1346 του 2000 και θα ήθελε να διατυπώσει η Νομική Επιτροπή ότι ο βασικός σκοπός του κανονισμού για τις πτωχεύσεις είναι να υπάρχουν κάποιοι κοινοί κανόνες όσον αφορά την ε, δικαστική ε, αρμοδιότητα ούτω ώστε να γίνει κάποια πτωχευτική διαδικασία και επομένως το εφαρμοστέο δίκαιο αφορά την αναγνώριση των ε, δικαστικών αποφάσεων όταν κάποιος οφειλέτης πτωχεύει. Αυτό όμως δεν σχετίζεται με δραστηριότητες κάποιων εταιριών όπως οι επιχειρήσεις που εδώ καταγγέλει ο αναφέρον. Επομένως, η αρμοδιότης να κρίνει ε, κανείς πότε μια μητρική εταιρεία όπως η μητρική εταιρεία της Πουέρτας Νόρμα προέβη σε απάτη ε, είναι αρμοδιότητα των τοπικών αργών. Ε, δηλαδή, σε αυτή την περίπτωση, των εθνικών δικαστηρίων. Ίσως είναι και αρμοδιότητες των περιφερειακών ή τοπικών αργών. Αυτά λέει η Νομική Επιτροπή, ότι αυτοί έχουν την, ε, την αρμοδιότητα της αξιολόγησης το αν υπάρχει απάτη ή όχι. Εν πάση είναι δικαστικό θέμα των εθνικών δικαστηρίων. Εμείς. <coughs> Στη συγκεκριμένη περίπτωση θεωρούμε ότι υπάρχει συμφωνία μεταξύ της μητρικής εταιρεία και των συνδικάτων που καλύπτουν τους εργαζόμενους αυτής της επιχείρησης. και το δικό σας συνδικάτο αλλά και τα άλλα ε, συμμετέσχουν στην σύνοψη αυτή της συμφωνίας. Στη συνέχεια τώρα ε, έχουν αναλυφθεί ενέργειες καταγγελίας στη δικαιοσύνη για αυτήν την απάτη που αφορά την αίτηση πτώχευσης. Είχαμε πέντε επενδυτές τελικά που ανέλαβαν την επιχείρηση αυτή από τις αρχές της Σόρια και το 2014 είχαμε την όρμα Doors Technologies η οποία ε, προσέλαβε 130 εργαζομένους της Πουέρτας Νόρμα. Πάντως πριν αποφασίσουμε οριστικά τι θα κάνουμε με, για αυτή την αναφορά, θα δώσω το λόγο στους ε, συναδέλφου που θέλουν το λόγο. Κυρία Αλμπιόλ, σα ευχαριστώ. Πρώτα πρώτα να ευχαριστήσω του αναφέροντες που παρίστανται στην συνεδρίασή μα. Νομίζω ότι εδώ έχουμε μια συγκεκριμένη περίπτωση που αφορά μια γενικότερη προβληματική. Όταν ένας όμιλο εταιριών χαράσει τέτοια στρατηγική για να κάνει πτώχευση και καθάριση σε μια θηγατρική και μετά μεταφέρει δραστηριότητα σε άλλη εταιρεία και λαμβάνονται διάφορα μέτρα μετά σε σχέση με την πτώχευση όπως η καθάριση τότε μιλάμε για κάποια δόλια πρακτική όπως έγινε προκειμένου αλλά, αλλά έχει γίνει και σε άλλες περιπτώσεις αυτό μας δείχνει για το ότι χρειάζεται να υπάρξει νομοθεσία η οποία να καλύψει αυτό το πρόβλημα. Νομίζω σε αυτή την περίπτωση αυτό το οποίο προκύπτει είναι ότι είναι προβληματική η νομοθεσία που διέπει την διασυνοριακή πτώχευση. Δεν περιέχει ο ε, ισχύων κανονισμός τέτοιες περιπτώσεις. Άρα χρειάζεται θέσπιση νομοθεσίας. Γι' αυτό σας λέω, η Επιτροπή μας θα πρέπει να διαβιβάσει την αναφορά στην Επιτροπή. Και με μια επιστολή μας ίσως να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να νομοθετήσει για αυτές τις περιπτώσεις γιατί είναι εδώ και θέμα της ε, κοινωνικής επιχειρηματικής ευθύνης. Επίσης η Επιτροπή Απασχόλησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρόκειται να συντάξει κάποια έκθεση για την εταιρική κοινωνική ευθύνη και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Άρα θα πρέπει και στην Επιτροπή Απασχόλησης να διαβάσουμε την αναφορά. Όλα όσα είπαν οι αναφέροντες θα πρέπει να έρθει αυτό το κενό του ισχυρού κανονισμού. Δεν καλύπτει όλε τι περιπτώσει. Και από πλευρά ευθύνη νομίζω ότι η Επιτροπή Απασχόληση θα πρέπει κάτι να κάνει. Ε, muchas gracias, señora Albiol, señora Ballina. Sí, bueno, anda. Η κυρία Βαλίνα. Συμφωνώ με όσα επίσης να σα πω από την ότι Έχουμε το πρώτο έχουμε τους συντρόφους που εδώ να μας παρουσιάσουν τι συμβαίνει και αυτό δείχνει το τι γίνεται με, την, με τον συνδικαλιστικό αγώνα. Ε, είναι μια, μια πάλι μακρόχρονη και δεν είναι μόνο θέμα του κλεισίματος του εργοστασίου, αλλά είναι το ότι οι άλλοι συνεχίζουν να εκμεταλλεύονται το δημόσιο χρήμα ε, και να δημιουργούν μια προβληματική περίπτωση σε όλη την επαρχία. Άρα θα πρέπει αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να το προσέξει. Είναι αυτό ακριβώ που λέγαμε. Θα πρέπει να γίνει αναθεώρηση της ε, εργατικής νομοθεσίας και αναθεώρηση των συνισχύουν για τα ευρωπαϊκά ταμεία. Γιατί έτσι απεριμώνεται η επαρχία και η Αλλά επίσης θα πρέπει να καλυφθούν και τα δικαιώματα των εργαζομένων τι γίνεται με τις ε, καταστάση επιχειρήσεων, γίνεται απερίμωση ε, και φτωχοποίηση της, της επαρχίας. Θα πρέπει επομένω όλα αυτά να τα προσέξει και η Επιτροπή Απασχόλησης. Να δούμε, έχουν γίνει βήματα πρόοδου σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσον αφορά την εταιρική και κοινωνική ευθύνη. Να εξεταστούν αυτά υπό το φως αυτής της αναφοράς. Άλλο ενδιαφέρον να γνωμοδοτήσουν ποιες είναι οι επιπτώσεις της έλλειψης εναρμόνισης στην Ευρώπη όσον αφορά τις μετεγκαταστάσεις στα πλαίσια των επιχειρηματικών ομίλων όπως έγινε εδώ με την Πουέρτας Νόρμα. Είναι πολύ σοβαρή αυτή η υπόθεση. Τα ακούσαμε αυτά σήμερα. Το τι γίνεται και με την επικουρικότητα. Ε, γιατί τα θέματα απασχόλησης είναι συνήθως συναρμοδιότητα Ευρώπης και Ευρωπαϊκών κρατών μελών. Άρα θα πρέπει να υπάρξει μια επιστολή ε, που να καλύπτει τις τόσες αναφορές που έχουμε συζητήσει για αυτά τα θέματα για τέτοιες εκαθαρίσεις, τέτοιες πτωχεύσεις. Δόλιες πτωχεύσεις. να δούμε αν θα πρέπει να συνεχιστεί η επικουρικότητα και τι θα γίνει με αυτές τις μητρικές εταιρείες που χειραγωγούν έτσι τους εργαζομένους ε, και εις βάρος αυτών με, με τέτοιου είδους πολιτική όσον αφορά τις θηγατρικές υπηρεσίες. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ για τόσο μας εξηγήσατε. Ε, λέει ε, θέλουμε κάτι να, να διευκρινίσουμε ότι δεν ζητούμε κυρώσεις εις βάρος της ε, πολυεθνικής. Ό,τι ήταν να κάνουν το κάνανε. Όμως σημαίνει το εξής, ότι έχουμε τώρα αυτή την εμπειρία. Η εμπειρία από αυτό που έγινε είναι το ότι υπάρχουν διάφορα κενά και αυτό θέλουμε ότι το 2002 σε σχέση με την ενάτη οδηγία για το δικαίωμα των εταιριών κατόπιν της έκδοσης Winter ε, είναι κάτι το οποίο δεν έλαβε συνέχεια. Θα πρέπει να εμβαθυνούμε σε αυτό γιατί είναι κάτι το οποίο αφορά την νομοθεσία στις χώρες προέλευσης αυτών των επιχειρηματικών ομίλων. Πρέπει να υπάρξει εναρμονισμένη ρύθμιση τα ισπανικά δικαστήρια έκριναν ότι πρόκειται περί απάτες. Γιατί διαπίστωσαν ότι γίνεται η πτώχευση, ζητείται η πτώχευση για να γίνει η μετεγκατάσταση. Άρα θα πρέπει να υπάρχει νομοθετική ρύθμιση για αυτές τις περιπτώσεις. Επομένως ο επόμενος κανονισμός για την εταιρική γεωνική ευθύνη πώς τη λέτε θα πρέπει κάτι να λέει όσον αφορά τέτοιες συμπεριφορές μητρικών εταιριών ή εταιρικών ομίλων, ιδίως όσον αφορά την ε, Ήπεθρο. Γιατί εδώ η πολυεθνική, η μητρική εταιρεία προκάλεσε κρίση, ε, έπληξε πάρα πολύ με αυτό το οποίο έγινε όλη αυτή την περιοχή, αυτή την επαρχία. Οπότε, τι να σας πω, επαφήμεθα στα όσα θα κάνετε εσείς. Ευχαριστούμε εμεί κύριε Ερνάντ, λέει πρόεδρο πέραν των όσων είπαν οι συνάδελφοι και εγώ θα πρέπει να επισημάνω ότι μου φαίνεται πάρα πολύ σημαντικό να εκμεταλλευτούμε αυτή την ευκαιρία γιατί που μας, που μας ε, ανέδειξε αυτή η έκθεση αυτή η ε, αναφορά για την κοινωνική εταιρική ευθύνη. Οι εταιρείε με σωστή συμπεριφορά θέλουν να υπάρχει υποχρεωτικά τέτοια κοινωνική ευθύνη. Τώρα, συμπεράσματα. Λάβουμε υπόψη τι είπαν οι συνάδελφοι. Και θα κρατήσουμε την αναφορά ανοιχτή. Όμως, ούτε η δική μας Επιτροπή μπορεί να προχωρήσει περαιτέρω αλλά θα ζητήσουμε και θα κάνουμε τις ενέργειες που είπαμε. Δηλαδή θα διαβιβάσουμε στην Επιτροπή Απασχόλησης την αναφορά για να ληφθεί υπόψη για την συντασσόμενη έκθεση. Χρήση, αξιοποίηση των κοινωνικών πόρων. Τι γίνεται με τα κοινωνικά ταμεία, όπως το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης. Τι γίνεται με τις επιπτώσεις των μετακαταστάσεων. Και πώς θα εφαρμοστεί την ε, απασχόληση η επικουρικότητα και κάπως να καλυφθεί η περίπτωση της δόλιας πτώχευσης και καθάρισης. Αυτά όλα να τα λέμε υπόψη για την έκθεσή τους. Αλλά και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ευάσουμε όλα τα στοιχεία. να ληφθεί υπόψη το τι είπε η νομική επιτροπή. Βέβαια την κυρίως αρμοδιότητα, γιατί τέλος την πιο αποφασιστική ενέργεια θα την κάνει η Επιτροπή Απασχόλησης. Τώρα έχουμε τη γνωμοδότηση της Νομικής Επιτροπής. Θα πρέπει να πούμε ότι η αρμοδιότητα για να γίνει η κρίση, η αξιολογική κρίση, εάν έχουμε εδώ ή όχι απάτη, αυτό είναι θέμα των εθνικών δικαστηρίων. Οπότε να στείλουμε και μια επιστολή στο Ισπανικό Υπουργείο Εργασίας, να ενημερωθούν για το τι γίνεται. Να ξέρουν ότι ξεκινάμε και συνεχίζουμε τη σχετική διαδικασία σε όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Να έχουν υπόψη τους επίσης το τι είπε η νομική επιτροπή. και να μας πούν αυτοί τι πιστεύουν. Κυρία Ελμπιόλα, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ. Ναι, ναι, συμφωνώ. Με τα συμπεράσματα. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να διαβαστεί το υλικό στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διαπίστωση του κενού κλπ. Δεν κατάλαβα το είπα αυτό. Ναι, ναι, δεν το, δεν το είπα ξεκάθαρα λέει πρόεδρο, αλλά και στην Επιτροπή Απασχόληση. Να ελάβει και η Επιτροπή Απασχόληση για την έκθεσή τη αυτά όλα. Αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν έγινε διαβούλευση, δεν ζητήθηκε η γνώμη της, με τη γνώμη της νομικής επιτροπής. Άρα και οι άλλοι να ενημερωθούν να ξέρουν τι αποφασίστηκε για το ποιος μπορεί να κάνει κάτι, τι γίνεται με τις τοπικές αρχές όπου θα πρέπει να ξέρουν τι γίνεται και θα ξέρει, να ξέρει επίσης και το Υπουργείο Απασχόλησης. Όλοι να ξέρουν την γνωμότητα της Νομικής Επιτροπής. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Ερνάντες. Ευχαριστούμε για όσα κάνατε. Έχετε κάτι να ερωτήσετε. Άρα, τελειώσαμε. Άρα, άλλη μία, άλλη μία είναι. Νομίζω τελειώσαμε σημερινή συνεδρίαση. Α, όχι, όχι, όχι. Πάμε τώρα στην τελευταία αναφορά. Αλλά βέβαια θα να σας ε, ευχαριστήσω για την συνεργασία σας, να σας αποχαιρετήσω και προχωρούμε. Uh, Κυρίες και κύριοι, έχουμε τελευταία αναφορά. 2669 του 2013 του Καρλ Μάιερ από τη Γερμανία για παραβίαση των βασικών διατάξεων του Δικαίου Ευρωπαϊκής Ενώσεως ας Γενικής Θήσης Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο αναφέρον απουσιάζει αλλά θα μας παρακολουθεί στο διαδίκτυο. Ας περάσουμε αμέσως στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριος Έρτινγκ λοιπόν έχει το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε το λόγο. Πράγματι είναι η περίπτωση Γερμανού αναφέροντας που μένει στη Γαλλική Πολυνησία και ζήτησε κοινωνική, ευεργετήματα κοινωνικά για ηλικιωμένου ότι την τοπική αυτοδίκηση του το αρνήθηκαν διότι θεωρήθηκε ότι δεν γεννήθηκε στη Γαλλική Πολυνησία και δεν ήταν Γάλλος να In this respect, the petitioner claims... Σχετικά με αυτό αναφέρον λέει ότι αυτή η άρνηση παραβιάζει τα δικαιώματά του σύμφωνα με Ευρωπαϊκή Σύμβαση για κοινωνική και ιατρική βοήθεια του 1953. Σχετικά με αυτό είχαμε πει ότι αυτή η σύμβαση δεν ε, αποτελεί τμήμα του ευρωπαϊκού δικαίου. Είναι μια σύμβαση που συνήθει υπό την αιγίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης Ιστρασβούργων και επιπλέον τα άλλα ευρωπαϊκά μέσα που αναφέρει δεν είναι εφαρμοστέα στη Γαλλική Πολυνησία, όμως επιμένει. Λέει ότι η Γαλλική Πολυνησία αποτελεί ένα στο τμήμα της Γαλλίας και η Γαλλία σίγουρα είναι κάτω μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, αδιαφυσβήτητα. Όμως, σχετικά με αυτό μπορούμε να επαναλάβουμε μόνο ότι η Γαλλική Πολυνησία είναι μέρος των μη ευρωπαϊκών χωρών και εδαφών που αναφέρονται στο παράρτημα 2 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα, συνεπάγεται και αντιστρόφως ότι είναι συνδεδεμένη με την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με το άρθρο 198 και 204 της συνθήκης. Άρα, δυστυχώς, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως δεν εφαρμόζεται αυτομάτως σε αυτά τα εδάφη ανεξάρτητα από το καθεστώς που απολαμβάνουν στην εσωτερική τάξη ενός κράτους μέλους, εν τη αυτή περιπτώσει της Γαλλίας. Και συνεφώ μπορούμε να διατηρήσουμε το συμπέρασμά μας ότι ο αναφέρον δεν μπορεί να επικαλεστεί ευρωπαϊκό δίκαιο ώστε να ε, ζητήσει τα ε, ευεργετήματα αυτά τα κοινωνικά ή στην γαλλική πολυνησία. Σα ευχαριστώ και τώρα να συζητήσουμε, να δώσουμε το λόγο στα μέλη. Θέλει κανεί να πάρει το λόγο? Όχι. Μάλιστα. Ακούσαμε την εξήγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και φαίνεται ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε. Γιατί αυτό δεν εμπίπτει στο ευρωπαϊκό δίκαιο, στην ευρωπαϊκή νομοθεσία και δυστυχώς νομίζω ότι είμαστε αναγκασμένοι να κλείσουμε την αναφορά αυτά. Αλλά η κυρία Πιτέρα θέλει το λόγο. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. εξ ονόματος του συναδέλφου που ασχολείται και με την ε, αναφορά αυτή και δεν μπορεί να είναι παρόν σήμερα, ήθελα να πω δύο λόγια. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω την πρότασή του. Η αναφορά αυτή να κλείσει. Γιατί προβλήθηκαν επιχειρήματα και αυτό θα επιτάσσαν τα επιχειρήματα τα οποία ακούσαμε Επίσης, ζητήθηκαν έγγραφα δικαιολογητικά, τα οποία δεν χορηγήθηκαν από τον ε, Ετούντα. Και έτσι λοιπόν πιστεύουμε ότι θα πρέπει να κλείσει η αναφορά. Μάλιστα, λέει ο Πρόεδρο, πιστεύω ότι θα πρέπει να κλείσει η αναφορά και να συστήσουμε στον αναφέροντα να υποβάλει ξεχωριστή αναφορά για το ζήτημα του Αμαζονίου. Αλλά αυτό δεν εμπίπτει στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας. Δεν μπορούμε λοιπόν παρά να σας συστήσουμε να τραφείτε σε άλλα όργανα. Μιας και αυτό δεν εμπίπτει στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Επιπλέον. Έγιναν κάποιες ερωτήσεις και αιτήματα για διαρευνητική αποστολή. Δυστυχώς ο κανονισμός προβλέπει ότι τέτοιες αποστολές διοργανώνται μόνο για εκκρεμείς αναφορές. Δεν μπορούμε να συζητήσουμε όμως περαιτέρω τη συγκεκριμένη αναφορά και ως εκ τούτου δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε και στο ετοιμά σα. Άρα θα πρέπει να κλείσει η αναφορά. Δεν βλέπω να υπάρχουν αντιρρήσει. Ευχόμαστε ό,τι καλύτερο βέβαια στον αναφέροντα και ελπίζουμε να κατανοείτε ότι έχουμε και δεσμευτικέ ε, διαδικασίε τις οποίες και πρέπει να τηρήσουμε. Μάλιστα, λοιπόν, ολοκληρώνεται λοιπόν το θέμα αυτό στην ημερήσια διάταξη. Και έτσι λοιπόν ολοκληρώνεται και η συνεδρία στη σημερινή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα λέμε την άλλη φορά.